Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να καθυστερήσω περισσότερο, αλλά έχουμε 43 σελίδες ψηφοφορίας τώρα. 43 πόσο θα καθυστερήσουμε ακόμα με το να μην μπορούμε να τακτοποιήσουμε στο σώμα εδώ τη διαδικασία ψηφοφορία. Είπαμε στην αρχή ότι θα αρχίσουμε στι 12, τώρα θα είναι μία παρα 10 και θα περάσει αρκετό χρόνο πρωτού τελειώσουμε. Σα καλώ να καλέσετε τον Πρόεδρο και το Προεδρείο για να διευκρινίσουν προ του επιτρόπους, Προεδρείο και άλλου να κινούνται γύρω από το δικό μας χρονοδιάγραμμα και να ψηφίσουμε εκεί που προβλέπετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι προβλεπόταν στις 12.30 η ώρα ψηφοφοριών. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση 20 λεπτών και όχι 40. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Φιντάντσα παντρεύτηκε και θα πρέπει να το συγχαρούμε. Και όπως είπατε, σήμερα προβλέπεται μία μακρά διαδικασία ψηφοφοριών με σωρία τροπολογιών, κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει δύο ώρες από τώρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να είμαστε γρήγοροι, αλλά θα πρέπει να μην διακυβεύσουμε τη σαφήνεια. Άρα βασίζομαι στη συνεργασία σας, διότι είναι μια μακρά διαδικασία και θα πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Περνάμε στην έκθεση ΕΚ, λοιπόν. Αρχίζουμε. Ψηφίζουμε με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. La relazione... Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Έκθεση των Εσόφσκι ζήτησε το λόγο, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη. Δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει κάποιος το λόγο. Εάν δεν το επιθυμείτε, ψηφίζουμε την έκθεση το Ζενόφσκι με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε την έκθεση Γκλάντε με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία συγχαρητήρια. Ε, έκθεση Ρόιλ. Ψηφίζουμε την έκθεση όχι με ονομαστική αλλά διανατάσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τσβιεύσκα. Τσιεύκα. Μπορεί να μιλήσει ο εισηγητής αν το επιθυμεί. Δεν το επιθυμεί. Α, επιθυμεί. Ναι, είναι δικαιωμάτο. Είναι δικαιωμάτο. Δεν μπορείτε να του το αρνηθείτε. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να καθιερώσουμε ένα μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Θέλω λοιπόν να πω ε, ότι κατέθεσε μια ενημερωτική, μια τροπολογία επικαιροποίησης. Μετά από την ψήφιση στην Νομική Επιτροπή 14 κράτη-μέλη που προσχώρησαν σε αυτό το μηχανισμό συμπεριλαμβανομένες και της Πορτογαλίας και της Μάλτας που είναι νέες χώρες. Γι' αυτό στο σημείο G πρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό από 12 σε 14. Και στη δεύτερη θέλω επίσης να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό ενισχυσμένης συνεργασία. Ε, να ευαισθητοποιήσουν για το μηχανισμό αυτό όλα τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο του 228 σημείο 1 της Συνθήκης για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω αυτός ο μηχανισμός να αποτελέσει ένα εργαλείο για την ε, καθιέρωση ειδικών δράσεων για περιορισμένο μόνο αριθμό χωρών. Ψηφίζουμε την έκθεση με ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε επίσης με συντριπτική πλειοψηφία. Έκθεση Σικλούνα ψηφίζουμε την έκθεση με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Σούριαν. Έκθεση Σούριαν. Να διευκρινίσω ότι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή 369 ψήφοι Ψηφίζουμε με ονομαστική την έκθεση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Σούριαν. Σαρνέτσκι. Θέλει ο εισηγητής το λόγο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι από αυτά που μας λέει το Συμβούλιο. Η συνεργασία ελπίζουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι υπήρξε μέχρι σήμερα. Ε, ποιοι είναι υπέρ της 33 κατά αποχές εγκρίνονται οι 33 τροπολογίες. 12, 46, 48. Υπέρ παρακαλώ. Αποχές εγκρίνονται. 13, 21, 29, 47. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20... 23 λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 23. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε να ελέγξουμε αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκανα λάθος εγώ, με συγχωρείτε. Αλλά δεν είναι της δικής μου ομάδας, δεν το έκανα σκόπιμα. Ψηφίζουμε την 24, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 3. 8 και 34 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 και 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 27 και 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 2 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος αρχίζει η ψυχοφορία πέρας εγκρίθηκε ψηφίζουμε τις 10 και 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Τροπολογίες 14 και 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Και εδώ θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 και 37 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 και 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 15 και 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 17 και 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 18 και 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 4 υπέρ. Έχετε το λόγο. ψηφίσουμε στη... για την απαλλαγή. Και θυμόσαστε ότι ψηφίσαμε και την προηγούμενη φορά. Και παρέμεινε ένας τίτλος λόγω της αναβολής της απαλλαγής. Θα ήθελα να διαγραφεί αυτός ο τίτλος καθώς και ο επόμενος. Λοιπά μέτρα και τεκμηρίωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λάθος. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η διόρθωση που θα έπρεπε να γίνει αυτόματα για να προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα. Δεκτών λοιπόν. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Με μεγάλη πλειοψηφία να συγχαρούμε τον εισηγητή. Έκθεση Λάντφορτ. Ψηφίζουμε το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 1 με ξεχωριστή ψηφοφορία. Αφορά την τροπολογία 1 και όχι την 10ε. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Το αντίστοιχο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής Αστροποποιήθηκε τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ε, σχέδιο ψηφίσματος ε, με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Έκθεση Bauer. Να εξετάσουμε την πρόταση οδηγίας. Έχουμε δύο αιτήματα πανομοιότυπα απόρριψης, ένα από την Επιτροπή Απασχόλησης και μία από κάποιους ε, ευρωβουλευτές υπό την ηγεσία του κυρίου Σούλτς. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική κλίση τις δύο προτάσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται οι προτάσεις. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχει ζητήσει το λόγο η συγγήτρια. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, πρέπει να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μάθουμε αν σκοπεύει να διατηρήσει την πρόταση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το Κολέγιο των Επιτρόπων θα εξετάσει τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές με ταξί αυτών και απόσυρση της προτάσεως μετά από την ψηφοφορία σας. Θα διαβουλευτούμε και με τις χώρες μέλη σχετικά με το πώς εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς και πώς συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις αυτές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Προτείνω λοιπόν να αναστείλουμε το θέμα αυτό βάσει του άρθρου 56. Κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την παρέμβαση του Επιτροπού αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται να αποσύρει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού την απορρίψαμε. Άρα τότε δεν χρειάζεται εκ νέου παραπομπή στην ε, Επιτροπή απασχόληση, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόληση. Εγώ από τα όσα είπε ο Επίτροπος, κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Εάν όντω ε, εγκριθεί, είναι προφανέ ότι έχετε δίκιο, κυρία Μπερέ. Εάν ο Επίτροπο επιβεβαιώσει ότι είναι διατεθειμένη να αποσύρει την πρόταση, είναι σαφέ ότι το Προεδρείο, το οποίο εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, δεν θα ξαναστείλει το θέμα στην ε, αρμόδια Επιτροπή. Αυτό θα κάνετε, κύριε Επίτροπε. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι είπα ότι το η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις εναλλακτικέ περιπτώσεις, καθώς και αυτήν που μας είπα. Κυρία Μπέρες. Κύριε Πρόεδρε, υπό τη αυτά συνθήκας και επειδή δεν είναι βέβαια τα πράγματα, από την απάντηση του Επιτρόπου ζητώ με βάση το 65.3 66.3 η Ολομέλεια να αποφανθεί επί του νομοθετικού ψηφίσματος που απορρίπτει την πρόταση της Κομισιόν και παρακαλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν το νομοθετικό ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Κυρία Μπερές, έχετε κάθε δικαίωμα φυσικά να το κάνετε αυτό. Έχει ζητήσει το λόγο η συγγήτρια τώρα. elnök úr, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a hogy Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων δεν είναι τεράστιος. Θα μπορούσε κανείς να προσφύγει κατά των 27 κρατών, αλλά δεν θέλω να συμβάλλω σε μια τέτοια προσπάθεια. Ωραία λοιπόν. Υπάρχει όμως η πρόταση της ε, Πρόεδρε τη Επιτροπή κυρία Μπερέ, θα ήθελα να ζητήσω κάποιον αγορητή υπέρ τη πρόταση και κάποιον κατά της πρόταση. Ποιο είναι κατά τη πρόταση κυρία Μπερέ, ε, για να ψηφίσουμε την ε, ε, πρόταση απόρριψη τη νομοθετικής πρόταση και ποιο Υπάρχει κάποιος κατά? Κανεί. Ωραία λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ? non c'entra niente. Non No, no, non è un problema di... Δεν ε, ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι. Βάσει του κανονισμού δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θεωρείται μη παραδεκτό το αίτημα της κυρίας ε, Περβάνς Μπερές. Μπορείτε να καθίσετε στις θέσεις σας. Η πρόταση τίθεται προς ψήφιση βάσει του κανονισμού. Πρόκειται για μια πρόταση την οποία θα ψηφίσουμε. Μπορεί να μιλήσει ένας συνάδελφος υπέρ και ένας κατά. Ποιο θέλει να μιλήσει υπέρ της πρότασης. Σε προηγούμενη περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, όταν είχε ψηφίσει για να απορρίψει πρόταση της Επιτροπής ε, και ήταν σχετικά με τα αποθέματα, αυτή η συγκεκριμένη πρόταση επανέκαμψε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή διότι δεν είχε πει θετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αποσύρει την πρότασή της. Εγώ θεωρώ ότι ο Επίτροπος επέλεξε πολύ προσεκτικά τις διατυπώσεις που χρησιμοποίησε και δεν συμφωνώ με την κυρία Μπερέ στην ερμηνεία που κάνει. Δεν θα γνωρίζουμε ακόμα εάν θα αποσύρει την πρότασή της ή όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς. Ο κύριος Τσίτσεστερ μίλησε κατά της πρότασης λοιπόν της κυρίας Μπερές. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Τούρμεν. Yes, I would like to speak in favor of Είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε τις ε, ψηφοφορίες μας σήμερα. Αναφέρομαι στο άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού. Εάν δεν αποσύρει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το Κοινοβούλιο παραπέμπει εκ νέου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρόταση για να υπάρξει νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα, εκτός εάν μετά από πρόταση της έδρας ή μετά από πρόταση πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 50 μελών συνεχίσει και ψηφίσει το σχέδιο ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό μας ζητήθηκε, είναι ξεκάθαρη η μετα απο προταση πολιτικης ομαδας η τουλαχιστον 50 μελων συνεχισει και ψηφισει το σχεδιο ψηφισματος νομοθετικου περιεχομενου αυτο μας ζητηθηκε ειναι ξεκαθαρη κατασταση ας προχωρήσουμε λοιπόν έτσι. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Επομένως, ψηφίζουμε την πρόταση να περάσει η πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Θέλετε διανατάσσεως χειρός? Διανατάσσεως χειρός. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Η πρόταση της κυρίας Μπερές εγκρίνεται. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Βόμποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να είχαμε δει διαφορετική εξέλιξη της ψηφοφορίας εάν η κυρία Συγήτρια είχε τηρήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και παρακαλώ στο μέλλον να γίνεται αυτό. E λοιπόν, συνάδελφοι, να ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ανοιχτή πέρασε της ψηφοφορίας. La risoluzione. Allora, abbiamo votato. Ψηφίσαμε λοιπόν για την απόρριψη της πρότασης νομοθετικού ψηφίσματος. Εγκρίνεται 383 ψήφοι υπέρ, 263 κατά. Επομένως, η έκθεση απορρίπτεται. Πέρα της διαδικασίας, προχωράμε. Έκθεση Σόμερ. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής Unblock. 155 τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. Η εισηγήτρια φυσικά μπορεί να παρουσιάσει την πρότασή της. Δεν θέλετε να παρουσιάσετε την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται μοναχά για μια ε, φραστική διευκρίνηση και μόνο για τα γερμανικά. Για τις υπόλοιπες μεταφράσεις δεν υπάρχει θέμα και το λέγω μόνο για ασφάλεια δικαίου. Διορθώνεται δηλαδή ο σωστός όρος των προσυσκευασμένων αυτών τροφίμων. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αντιρρήσεις με αυτή την τροπολογία. Συναδελφοί, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη βούλησή σας, αλλά πρόκειται για μια τροπολογία η οποία αφορά απλώς την γλωσσική γερμανική εκδοχή. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό να είναι κάποιος αντίθετος ε, για μια τροπολογία η οποία δεν έχει να κάνει με την ουσία της ε, υπόθεσης. Βέβαια είναι δικαίωμα του καθενός να ε, είναι αντίθετος και να εκφράσει τις αισθάσεις του. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποσύρετε αυτή την ένσταση. Εγκρίνεται λοιπόν η προφορική τροπολογία και υποβάλλεται προς ψήφιση μαζί με την τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά να κάνουμε έναν έλεγχο για την τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 48. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Η τροπολογία 50 εγκρίνεται. Προφανώς δεν σηκώσετε τα χέρια σας όταν ψηφίζαμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά την επόμενη φορά, δηλαδή τώρα, να σηκώνετε το χέρι σας. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εμένα μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Αν θέλετε να το, εγκρίνουμε, ε, να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά, να κάνουμε έναν έλεγχο. Σφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. να κάνουμε έναν έλεγχο. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 124. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 130. Με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Θέλετε να την παρουσιάσετε. Κυρία Σόμερ, παρακαλώ. Ε, Στην προκείμενη ε, τροπολογία μάλλον, πρόκειται για την επαϊσίμαση τροφίμων που περιέχουν νανοτεχνολογικό υλικό. Εφόσον πρόκειται για στέρεο νάνο υλικό, γιατί υπάρχει και το μη στερεό. Για παράδειγμα, ζάχαρη η οποία έχει αλεστεί τόσο πολύ ώστε έχει φτάσει πλέον να είναι σε επίπεδο μεγέθους νάνο η ζάχαρη αυτή, η οποία όμως δεν ε, επηρεάζει καθόλου τον οργανισμό. Μιλούμε λοιπόν για στέρεο ε, ή σταθερό υλικό. Υπάρχουν ενστάσεις. Επειδή Έχουμε πάνω από 40 συναδέλφους που είναι κατά. Η προφορική τροπολογία δεν γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 130. Υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Τροπολογία 131. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασης ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να κάνουμε παλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές φαίνεται ότι απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εμενταμέντο 210. Τροπολογία 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 232 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 244. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 286. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Τροπολογία 39. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 292. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 350. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 293 με ονομαστική κλίση. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. τεράστια πλειοψηφία. Τροπολογία 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρασε η ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Συγγνώμη. Τροπολογία 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 326. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 284 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Τροπολογία 87 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 326 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 257 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση στην τροπολογία 251. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. με ονομαστική κλίση τη 252. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώνεται την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 253 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ο κύριος Βίλμοντ ζητά να προτείνει, η κυρία Βίλμοτ ζητά να προτείνει μια προφορική τροπολογία. Τη δίνουμε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να αλλάξει λίγο η παραγραφό, να λέει δηλαδή ο τόπο προέλευση. Θα είναι τότε νομίζω διαφανέστερο για του καταναλωτέ. Υπάρχουν ενστάσεις. Eh, Και εδώ πραγματικά μου φαίνεται λίγο υπερβολικό να είμαστε αντίθετοι σε μία γλωσσική αλλαγή. Τώρα προέλευση, καταγωγή, σιγά τη διαφορά. Αλλά αν υπάρχουν στάσεις δεν μπορώ να δεχτώ την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε κατά τμήματα λοιπόν. Τροπολογία 101. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Με ονομαστική κλίση, ζητώ συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα και πάλι με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 254. Υπέρ, κατά, αποχές, ελάχιστε ουσίδα. Ξανακάνουμε, επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Υπέρ. Η εισηγήτρια ζητάει το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο τμήμα της 101 εγκρίθηκε, το δεύτερο απορρίφθηκε. Κατά την κρίση μου πρέπει να πάρουμε από την τροπολογία 328. Αυτήν πρέπει να την υπερψηφίσουμε. Πρόκειται για την τεχνική προσαρμογή στα πλαίσια της προσαρμογής που κάνουμε μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας και την θέση της εφαρμογή εκεί πρέπει να περιληφθεί ο όρος delegated, delegated act αντί για την διαδικασία της επιτροπολογίας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ψηφιστεί αυτή. Έχετε δίκιο κυρία Σόμερ. Ωραία. Να ψηφίσουμε εκ νέου την τροπολογία 328 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 254. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 333 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 334 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γερμανικά, κύριε Σούλτς. Αν μου τα πείτε ιταλικά, έχει καλός. βιάζομαι κύριε Σούλτς, γι' αυτό υποβάλλουμε προς ψήφιση την 311 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 267 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 324 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 121 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος είναι υπέρ για την 121 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 125 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 127. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 264 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 294 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 336. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 259, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 337, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 338 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 268 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 295 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Mm-hmm. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τροπολογία αυτή δεν μιλάει καθόλου για τα For four should still be voted. για τα trans fat, για τα λιπίδια αυτά, αυτού του είδους. Διότι είναι σημαντικό θέμα για πολλούς από εμά εδώ. για τα υπερλιπίδια. Κυρία Χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία του θέματος και να κάνω συζήτηση, είναι μια λύση που δόθηκε από το λεγόμενο Tabling Office, όπως αναφέρεται αυτή στην λίστα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζητεί διαγραφή του άρθρου 29 11β. Αυτά που εννοεί ο κύριος Σλούτερ είναι πράγματα τα οποία μπήκαν ως Β στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά έχουν την αρρύθμιση ΒΑ. Γι' αυτό θεωρεί ο κύριος Λούιτερ ότι αυτή η προσθήκη πρέπει να γίνει στο 2911Β και επομένως είναι έξτρα προσθήκη και δεν συμπίπτει με τη νέα τροπολογία για την παράγραφο αυτή που βρίσκεται στον κατάλογο ψηφοφορία σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η λύση που έδωσε το Tabling Office και θα πρέπει να εκπίπτει 144 εάν εγκριθεί η 295. Επειδή όμως υπάρχει απόκληση απόψεων και επειδή πρέπει να πω ότι ο κύριος Σλίτερ είχε και την εντιμότητα να με ενημερώσει πριν να υποβάλει το αίτημά του αυτό στην Ολομέλεια, γι' αυτό προτείνω να ψηφίσουμε έξτρα την 144. Διακόπτη το μικρόφωνο. Allora, onorevole Sommer. Κυρία Σόμερ, πέστε μας, αν έχει δίκιο ο κύριος Σίλτερ. Δεν έχει δίκιο, οπότε ψηφίζουμε τη 295 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. L'abbiamo già fatto. Άλλο... Την έχουμε ήδη ψηφίσει, επομένως, πίπτη 144. La votazione è chiusa. Πέρασε της ψηφοφορίας. Η τροπολογία απορρίπτεται. Επομένως, ψηφίζουμε την 144. La votazione... Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione... Πέραση ψηφοφορία. Η 144 εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δημιουργήθηκε μια κάποια σύγχυση. λόγω κάποιων εξωτερικών παρεμβάσεων. Τροπολογία 312 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση L'emendamento Απορρίπτεται. Πριν από αυτή την τροπολογία έπρεπε να ψηφίσουμε την τροπολογία 269 την οποία υποβάλλω τώρα προς ψήφιση. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται η τροπολογία και κατόπιν την 145 υπέρ. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε μια παλήθευση γιατί δεν έχουμε ανάταση χειρός. Η συγγήτρια παρακαλώ. Πρέπει να ψηφίσουμε την 339. Πάλι πρόκειται για τεχνική προσαρμογή και πρέπει να λέει πράξη κατεξουσιοδότηση. Delegated Act. Έχετε δίκιο, κύριε Συγήτρια. Ψηφίζουμε την 339 υπέρ. Κατά απόχέ συγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 340. Υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 341 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 313 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 313 από τρεις πολιτικές ομάδες, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, πάντα με ονομαστική κλίση. Κυρία Σόμερ. Έχει αποσυρθεί 313 και πρέπει επομένως να ψηφιστεί 149. Ψηφίζουμε την 149 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 313 πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 316 καταπίπτει. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. «297 με ονομαστική κλίση». Κύριο Σίλτερ, παρακαλώ. Λοιπόν, για το 31 υπεδάφιο 3. Το ΕΛΚ θέλει να διαγραφούν οι υποχρεωτικές ρήτρε που αναφέρονται εδώ και ο συντάκτης είναι υπέρ της 314. Αποφάσισε το 31 3α καινούριο να παρισφρήσει εδώ και άρα αν εγκριθεί η 297 καταπίπτει αυτή. Μα εσείς ε, δικάζετε τις προθέσεις. Πρώτα θα ψηφίσουμε και μετά θα δούμε τι πρόθεση υπήρχε. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 297 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 314 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασες τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 151. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 298 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 299 υπέρ κατά, αποχές, εκρίνεται. Τροπολογία 315 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 316 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. La τη Εγκρίνεται. Η εισηγήτρια, παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κανονικά δεν έπρεπε να ψηφιστεί η 316 γιατί εκπίπτει η 316 εφόσον εγκρίθηκε η 313. Η 313 χωρίστηκε σε δύο τμήματα, ψηφίστηκε δηλαδή σε δύο τμήματα. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πολύ, απορρίφθηκε, λάθος έκανα. volta Ε, πότε εμεί, πότε εσεί, όλο και κάποιο λαθάκι κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Για να υπάρχει ισορροπία. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού τις τροπολογίες 158 και 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 300 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 342 καταπίπτη και η 166. Τροπολογία 171 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 270 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 274 λοιπόν. Τροπολογία 301 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Votazione Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τραπολογία 346. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 347. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 348. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 349. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 191. Η εισηγήτρια, παρακαλώ, κυρία Σόμερ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε μόλις ότι απορρίφθηκε η 346. Νομίζω ήταν εσφαλμένη η κρίση σας. Πάλι εδώ πρόκειται για θέμα τεχνικής προσαρμογής και οι πολιτικές ομάδες έχουν συμφωνήσει. Παρακαλώ να επαναλάβετε. 346. Facciamo votare 346. Να ψηφίσουμε την 346, να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. 346. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ε, ναι. Εγκρίνεται η τροπολογία. Ε, άμα δεν σηκώνετε τα χέρια σας, εντάξει, καταλαβαίνω, κουραστήκατε, δουλεύουμε όλη μέρα, αλλά άμα δεν σηκώνετε τα χέρια σας, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι θέλετε. Ψηφίζουμε την 191 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione. Πέρασε ψηφοφορία. L'emendamento ha ottenuto gli Απορρίπτεται 309 υπέρ 309 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 302 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 322 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 304 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 317 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 275 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 276 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 262 και 321 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 219 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 302 υπέρ, 305 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 229 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 263 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 278 καταπίπτει. 279 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 280 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 236 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 281 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 307 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 256 υπέρ. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 323 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 282 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία για την 318. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Ψηφίζουμε τις 246 και 247 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 319 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 319. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τραπολογία 285 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 308. 308 υπέρ. Υπέρ της 308. Ποιος είναι υπέρ της 308. Κατά. Ρωτάω, ποιος είναι υπέρ της 308. Κατά. να κάνουμε την ηλεκτρονική υπαλήθευση για τη 285. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 309 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 329 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 330 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 331 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 332 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Ψηφίζουμε Μισό λεπτό. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Και εδώ έχουμε αθρώα πλειοψηφία. Να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, λόγω της προκεχωρημένης ώρας Παρακαλώ να ψηφίσουμε μόνο ακόμη τη 220 και την οικονομική διακυβέρνηση, τα υπόλοιπα δε αύριο. Και αν δεν αρκέσει και Παρασκευή πρωί. Υπάρχουν ενστάσεις για την πρόταση του κυρίου Ντόλ. Αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, ε, δέχομαι πολύ ευχαρίστως και γιατί θεωρώ ότι αυτά τα δύο θέματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε πολιτικό επίπεδο. Ξεκινάμε λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Ψηφίζουμε την παράγραφο 3 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Με αθρώα πλειοψηφία εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος. Συγχαρητήρια στους συντάκτες και στο Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Περνάμε τώρα στην οικονομική διακυβέρνηση. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Δεν είναι μονομαστική κλίση, υπέρ λοιπόν. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 31, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα μονομαστική κλίση. Όχι. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με αθρώα πλειοψηφία. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα ήθελα τώρα να προτείνω να ψηφίσουμε και την Ειδική Επιτροπή για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Πρόκειται για μία απλή ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έχουμε και την αντιπροσωπεία Καριφόρουμ με την πρόταση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη σε όλους.